Good morning, dear colleagues. Um, Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, είναι και 8 και 6 και επειδή η συνεδρίαση είναι μόνο μία ώρα και πρέπει να τελειώσουμε ακριβώς στις 9, ε, ας αρχίσουμε. Έχουμε λοιπόν μια κοινή συνεδρίαση το πρωί για το σημείο 2 για την υπόθεση της νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε, το ξέπλυμα κοινό και το σημείο 3 συζήτηση για την κατεξοδότηση πράξη για την ταυτοποίηση ε, τρίτων χωρών ε, υψηλού κινδύνου. Έχουμε μέχρι 16 ομιλητές, δύο συνεισηγητές και 7 ε, σκιώδεις, επί 2, ένας από κάθε επιτροπή ε, τρίλεπτο ο καθένας και επειδή δεν έχουμε μία ώρα αλλά 51 λεπτά Ε, ε, παρακαλώ, οι σκιοδησηγητές τρία λεπτά, πέντε λεπτά οι συνεισηγητές. Η τέταρτη οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλήματος εγκρίθηκε στις 20 Μαΐου του 2015 στο πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση τρομοκρατίας το Φλεβάρι του 2016 κάλεσε τα κράτη-μέλη να ε, θα ανακοινώσουν μέχρι το τέλος του 2016 πότε θα μεταφέρουν την οδηγία. Έγιναν κάποιες τροπολογίες τον Ιούλιο που αφορούν θέματα διαφάνειας και χρηματοδότησης στα πλαίσια της κείμενης οδηγίας. Εγκρίθηκε λοιπόν ο πρώτος κανονισμός στην τέταρτη οδηγία με κατάλογο χωρών που έχουν στρατηγικές αδυναμίες, deficiencies, δύσκολη λέξη για Γερμανό να την προφέρει, και για την καταπολέμηση του ξεπλήματος. Ε, μια ενημερωμένη έκθεση, μάλλον ε, έκδοση του καταλόγου προτείνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 24 του μηνός και δεν θα ε, συμπεριλαμβάνεται το θέμα αυτό ε, ε, ε, συζητείται σήμερα και αν συζητήσουν, αν θεωρήσουν σκόπιμο τα μέλη της ΕΚΟΝ και της ΛΥΒΗ μπορεί και να απορρίψουμε την πρόταση. η Γκου έκανε ένα ψήφισμα στις 29 Νοεμβρίου άρχισε η γραπτή διαδικασία μεταξύ των συντονιστών η προθεσμία μετά τη σημερινή συνεδρία στις 12 για να δούμε τι θα αποφασίσουμε. Starting with um, the discussion, I would hand over to... Λοιπόν, θα παραδώσω τώρα στον πρόεδρο Μωράες, γιατί ξέρετε ότι είναι κοινή συνεδρίαση, ε, Λίμπε και ΕΚΟΝ. Εγώ ξεκίνησα, συνεχίζει Λίμπε, γιατί μοιραζόμαστε τη δουλειά και έχουμε 49 λεπτά. To use the time Uh, καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα το χρόνο. Θα ήθελα να προλάβουμε να ακούσουμε όλους, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Και θα έχουμε λοιπόν ε, ισχυώδεις εισηγητές και θα πηγαίνουμε ένας ένας, ένας έκον, ένας λίμπε και ούτω καθεξής. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Κάριντς που είναι ο, προ... ο εισηγητής ε, του... Ε, της ΕΚΟΝ. Πέντε λεπτά. Και ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Πάντοτε είναι ευχάριστο να ξεκινάμε νωρίς. Τώρα, όσον αφορά την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και του οικονομικού εγκλήματο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ο αγώνα συνεχίζεται. Πρέπει να ε, ξεκαθαρίσουμε ε, και να φωτίσουμε πολλά στοιχεία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας μετά τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι. Ξέρουμε ότι οι ανώνυμες κάρτες ε, χρειάζεται να ρυθμιστούν καλύτερα και μετά από τα Panama Leaks Επίσης δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για παράνομους σκοπούς που επίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Η κυρία Ζαργεντίνη που θα μιλήσει αμέσω μετά από μένα και θα πει αυτά που ξεχνάω, ελπίζω. Και ελπίζω ότι δεν θα φέρει αντιρρήσεις αυτά που λέω. Την τελευταία φορά που δουλέψαμε μαζί γι' αυτό το, το θέμα, ε, που συνεργαστήκαμε, ε, καταλήξαμε στα κύρια σημεία όσον αφορά τη ε, Μητρώα Ιδιοκτησίας. Θα μπορούσαμε να στρίξουμε τη δημόσια πρόσβαση σε αυτά και μάλιστα την τελευταία φορά είχαμε ε, μακρά συζήτηση για αυτό το θέμα, ενώ τώρα προτείνω συμφωνία με την Κομισιόν να ε, επικρατήσει εμπιστοσύνη όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Την άλλη φορά, ε, την περασμένη φορά, μάλλον φέρασε καθόλου από το Συμβούλιο. Βεβαίω, Εξαιρέσει θα υπάρξουν και θα γίνει και συζήτηση για το πώς θα ενταχθούν οι όμιλοι εδώ, γιατί βέβαια οι νόμιμοι όμιλοι έχουν μεγάλο ρόλο ειδικά σε μερικά κράτη-μέλη, σε ορισμένα κράτη-μέλη. Τέλος, Επόμενο σημείο. Ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες. Θα μειωθεί το όριο προβλέπουμε ότι οι ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στο ίντερνετ γιατί υπάρχει στοιχείο ανιχνευσιμότητας για αυτές τις κάρτες. Ίσως να μην είναι το χειρότερο αυτό το στοιχείο, αλλά θα μειωθεί το ε, όριο. Αν ακούσετε την Europol έχει μια άποψη, αν ακούσετε τους επιχειρηματίες η δική τους άποψη κάπως διαφέρει. Οπότε προσπαθούμε πάντοτε να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της καταπολέμησης του εγκλήματος χωρίς να πνίξουμε τις επιχειρήσεις αυξημένη συνεργασία. Υπάρχει έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Έχουμε κάποιες προτάσεις για να προσπαθήσουμε αυτό να το διορθώσουμε και η Κομισιόν προτείνει να δημιουργήσουμε όχι μόνο ένα μητρό των ε, ιδιοκτητών δικαιούχων αλλά και, και ένα μητρό τραπεζικών λογαριασμών. Συμφωνήσαμε ότι αν το έχουμε αυτό θα άξιζε να έχουμε και πληροφορίες για το ποιος έχει και θηρίδες. Εντάξει, χωρί, απόρριτο το τι έχει μέσα, τι είδους συναλλαγές ε, ε γίνονται στους τραπεζικούς λογαριασμού, απλώς ποιος έχει τι. Οπότε αν γίνεται μια έρευνα για σοβαρό έγκλημα, θα ε, ε, μπορεί να οι ερευνητέ να πάρουν τις ε, πληροφορίες. Ευχαριστώ, σταματώ. 3 λεπτά 25 και τώρα η κυρία Σαργεντίνου που είναι η για αυτό το θέμα στη ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα ξανά. Πριν τα Χριστούγεννα του 2014 δεν απατώμε, είχαμε τελειώσει την προηγούμενη προσπάθεια. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί η οδηγία αυτή και ειδού που βρισκόμαστε. Προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε μετά τις μεγάλες αλλαγές που έχουν επελθεί στον κόσμο. Σε ό,τι αφορά τι τρομοκρατικέ επιθέσεις ε, στο Παρίσι, μετά ακολούθησαν και τα έγγραφα του Παναμά Προσπαθούμε να φέρουμε διαφάνεια στο θέμα. Ήταν μια πολύ δύσκολη μάχη. Τώρα βλέπουμε και την Κομισιόν και το Συμβούλιο να ε, εστερνίζονται την ιδέα της διαφάνειας ε, για να αντιμετωπίσουμε τις παράνομες ροές κεφαλαίων. Εγώ το βλέπω από τη σκοπιά της ανάπτυξης και θα πρέπει οι φόροι να πληρώνονται εκεί που παράγονται κέρδη. Βλέπουμε πάρα πολλά χρήματα να φεύγουν από μια ήπειρο όπως είναι η Αφρική αντί να επενδύονται και να ευημερεί ο κόσμος. Δύο νομοθετήματα έχουμε, την AMOD 5 και την ε, ε, οδηγία για το δίκαιο των επιχειρήσεων. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετέφερε το θέμα από την πρώτη οδηγία στη δεύτερη, όπου υπάρχει πρόσβαση χωρίς να πρέπει να δικαιολογείται το θεμητό συμφέρον καταλαβαίνουμε τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το σκεπτικό, αλλά ε, ε, εξαιρούνται τα ιδρύματα, ε, τα γερμανικά Stiftungen, όλα τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και δεν είναι εταιρείε, εξαιρούνται από το Δημόσιο Μητρό. Εμείς δεν θέλουμε να τα δούμε αυτά. Θέλουμε να ξαναμπεί στο AMLD4 και αυτό έχει σχέση με πολλές από τις τροπολογίες που έχει τις χέρια σας. Και επίσης θέλουμε να ενισχύσουμε ε, την ε, διατύπωση για τα trust, ε, για να εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται. Δεν θα πρέπει να έχουμε συστήματα στην Ευρώπη με εταιρείε θηρίδες ή εικονικές. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, παντού υπάρχουν τέτοια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τα trust με μια πάρα πολύ ευρία έννοια ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν ε, κάποια τραστ, κάποια καρτέλα, ακόμα και τα ονομάζουν διαφορετικά στην επικράτειά τους. Είναι καλός αυτός ο τρόπος που προτείνεται για να προχωρήσουμε. Ο κύριος Κάρινς μίλησε κάτι για τις προπληρωμένες ε, χρεωστικές κάρτες που είναι ανώνυμες. Αλλά υπάρχουν και γνωστές ε, δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πάρα πολύ αυστηρή διαδικασία για προπληρωμένες ε, χρεωστικές κάρτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς τα κατανοούμε όλα αυτά, αλλά υπάρχουν πολύ σκληρές ε, προϋποθέσεις και περιορισμοί για τις επιγραμμικές πληρωμές. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι εκτός ε, του κανονικού τραπεζικού τομέα και δεν μπορούν να κάνουν τις πράξεις τους και τις συναλλαγές τους ε, στο διαδίκτυο αν είναι τόσο στενός ο κορσές. Λοιπόν, βλέπουμε κάποιες χώρες να κάνουν κάποιες προσπάθειες και πολύ μεγάλες, ενώ κάποιες άλλες ε, δεν βιάζονται να μεταφέρουν στην νομοθεσία την οδηγία, γιατί οδηγία είναι και εμείς δεν έχουμε κανένα μέσο να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να το κάνουν. Εμείς ε, προσπαθούμε να τους πιέσουμε και παρακαλώ τους και σας, ε, σας έρθει καμία φαϊνή ιδέα να μας την πείτε. Ε, είναι προφανές ότι για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα θα πρέπει να την εφαρμόσουν την οδηγία όλα τα κράτη-μέλη. Έρχομαι τώρα στην κατεξοδότηση πράξη. Στείλαμε επιστολή στην Επίτροπο Γιούροβα ε, με την υπογραφή των Προέδρων Έκων και Λίμπε και των ε, συνσηγητών, υπογράψαμε και ο κύριος Κάρης και εγώ το Σεπτέμβριο, είπαμε ότι μας έχει κάπως απογοητεύσει ο κατάλογος των τρίτων χώρων που προτείνεται, ε, γιατί είναι ε, η λίστα του FATF ενώ ε, χρειάζεται στην οδηγία αυτή ένα κίνδυνο που θα τον έχουμε εκτιμήσει οι ίδιοι και όχι να αντιγράφουμε λίστες. Περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας φέρει ένα πιο φιλόδοξο κατάλογο μόλις ολοκληρωθεί η κατεξοδότηση πράξη. Τώρα δηλαδή. Δεν μας απάντησε επί της ουσίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη βλέπουμε τώρα ένα νέο κατάλογο που έχουν βγάλει μία χώρα. Δηλαδή αντιγράψανε το FATF. Από πλευράς των Πρασίνων ε, συμφωνούμε με την πρόταση της ΓΚΟΕ να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Την περασμένη φορά προσκαλέσαμε φιλικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση. Τώρα στο ψήφισμα μπορούμε να πούμε ότι ε, δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Τζούντιθ. Ο Πίτερ Σάιμον τώρα είναι ο συγητής της ΕΚΟΝ από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολλά βασικά σημεία που ζητούσαν οι σοσιαλιστές και δημοκράτες έχουν συμπεριληφθεί. Το είχαμε πει την περασμένη φορά ε, όταν μιλούσαμε για την τέταρτη οδηγία για το ξέπλυμα. Όλα αυτά που ζητήσαμε και το σχέδιο έκθεσης πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω τα έγγραφα του Παναμά ε, μας έδειξαν με τρόπο εντυπωσιακό πόσο ανάγκη υπάρχει για να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες οι εταιρείε για την καταπολέμηση του ξεπλήματος. Ε, λεπτομέρειες. Ποιος είναι ο οικονομικός ε, δικαιούχος τώρα. Υπάρχουν κανονικές εταιρείες και υπαθητικές ε, μη χρηματοοικονομικές. Τι θα πει αυτό. Ε, δεν υπάρχει τέτοια διαφορά, ε, δημιουργούνται παραθυράκια και τίποτα άλλο. Θα πρέπει να υπάρχει όριο για όλες τις ε, εταιρείες 10% του μετοχικού κεφαλαίου για το οικονομικό συμφέρον. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που ε, οι συγητές ασχολούνται και με ένα άλλο παραθυράκι θα πρέπει να αναφέρονται στο Μητρό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διαφάνεια. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση τώρα στο Κεντρικό Μητρό, καλωσορίζω επίσης τη δικτύωση των Κεντρικών ε, Μητρών και την ε, πρόσβαση του κοινού. Είναι σημαντικό αυτό γιατί δεν γνωρίζουν σύνορα η τρομοκρατία ούτε το ξέπλυμα χρήματος. Αλλά δεν μας βοηθάει ένα μητρό όσο καλό και να είναι, αν δεν βεβαιωνόμαστε ότι ε, ε όλες ε, οι ε, αρχές έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Για όλους τους υπολείπους που θέλουν να έχουν πρόσβαση στον κατάλογο, μπορούμε να επιβάλλουμε κάποιο διοικητικό τέλος. Ε, οι ε, διοκτικές αρχές τύπου ΣΔΟΕ και οι κρατικές αρχές θα πρέπει να έχουν δωρεάν πρόσβαση. Οι λοιποί να πληρώνουν ένα μικρό τέλος. Για τα τρας τώρα. Καλώς ορίζουμε επίσης τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και την τροπολογία 29 του σχεδίου έκθεσης. Σε ό,τι αφορά ε, τα κτηματολόγια, δηλαδή ε, την τροπολογία 33. Υποστηρίζουμε και την ιδέα αυτή, γιατί προσφέρονται φυσικά πάρα πολύ ωραία τα ακίνητα για θολές σκοτεινές συναλλαγές και για ξέπλυμα χρήματος. Αλλά και εδώ θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους τα κτηματολόγια. Ένα τελευταίο θέμα που το συζητήσαμε και την περασμένη φορά για την ε, νομοθετική διαδικασία για την τέταρτη οδηγία για το ξέπλυμα και με ενδιαφέρε πάρα πολύ ανέκαθεν, αλλά με μηδενική ε, επιτυχία έχω πει τα δημόσια πρόσωπα να μην είναι μόνο πολιτικοί και θα ξαναφέρω τροπολογία. Υπάρχουν ομάδες υψηλού κινδύνου όπως οι θύνοντες, ε, από την οικονομία, από τον αθλητισμό, ε, από τις εκκλησίες. Κοιτάξτε τι έγινε με το σκάδαλο FIFA. Τα δημόσια πρόσωπα που είναι εκτεθειμένα δεν είναι μόνο πολιτικοί, ε, είναι και άλλοι επιρρεπείς σε τέτοια πράγματα. Επίσης, ο, ο, ο κατάλογος αυτός, η μαύρη λίστα, είναι απαράδεκτος παίρνουμε ένα κατάλογο όπως έχει και βγάζουμε τη Βόρεια Κορέα και πάνω μας. Ευχαριστούμε, Πίτερ. Η Άννα Γκόμες είναι η επόμενη εισηγήτρια. Εγώ υποστηρίζω τους ΙΤΕΣ ως επιτοπλίστων και κυρίως αυτά τα περί καταπιστευμάτων που είπε ο κύριος Κάρης και για το Μητρό των Τραπεζικών Λογαριασμών. Νομίζω το είπε η Τζούντις αυτό, σε Αργεντίνη. Δεν είναι μόνο οι τραπεζικοί λογαριασμοί από ό,τι μαθαίνω για το ξέπλυμα μεγάλων ποσών χρησιμοποιούν συμμετοχή στις τράπεζες. Οι φίλοι από την ΕΚΟΝ νομίζω ότι θα έπρεπε να αποδώσουν τη δέουσα προσοχή σε αυτό το φαινόμενο. Ε, τώρα, η διεύρυνση του πεδίου για τις οντότητες ε, για να καλύψουμε και αυτούς που κάνουν consulting για φορολογικά ζητήματα ή για αυτούς ε, που κάνουν εμπορέο πολιτιστικών αγαθών, δημοπρασίες, τα, τα free ports όπου ατελώς ε, γίνονται συναλλαγές ε, με διάφορα πολιτιστικά αγάθα. Επίσης, ε, όσοι έχουν συμμετοχή πάνω το 10% σε οποιαδήποτε οντότητα. Οι, τα ανώτερα στελέχη που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ε, δικαιούχοι όταν δεν μπορούμε να βρούμε άλλους. Βάσει σύσταση ΓΑΦΗ, ε, γιατί το είπε και η Επίτροπο Γιούροβα σε μια απάντηση που μου έστειλε για ε, σε μια πρόσφατη ακρόαση της Επιτροπής ε, για το σκάνδαλο Παναμά. Νομίζω ότι ε, είναι αστείο διότι επειδή υπάρχει αυτό το παραθυράκι ε, θησαυρίζουν οι εγχώροι φορολογική παράδειση. Όποιο δεν ξέρει τον ε, δικαιούχο δεν μπορεί να, να αναλάβει μέτρα δέουσα επιμελητία. Οπότε ε, θα πρέπει να διακοπεί αυτή η ε, επιχειρηματική σχέση και για το Μητρό. Δεν είναι περίεργο που ο εκπρόσωπος νομικής εντότητας καταχωρίζει μια εταιρεία αλλά αρνείται να δώσει την ταυτότητα του δικαιούχου στο Μητρό. Είναι τεράστιο αυτό το παράθυρο που έχουμε ανοίξει ε, και δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται ε, κάτι τέτοιο στα Μητρέα. Ε, για τη διεύρυνση των κριτηρίων που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποτιμήσει αν η μία, χώρα, μία τρίτη χώρα είναι υψηλού κινδύνου προτείνουμε ένα κατάλογο πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων που πρέπει να εκπονείται και να επικαιροποιείται από τα κράτη-μέλη και μετά θα πρέπει να συλλέγει τις λίστες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι γελίο να ε, αγοράζουν υπηρεσίες από αναξιόπιστες αμερικανικές ε, εταιρείες. Ε, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό κατάλογο δημόσια εκτεθειμένων προσώπων και το κεντρικό Μήτρο Επιχειρήσεων και Τρας όπως είπα, το Μητρό πρέπει να καλύπτει και οντότητε που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανοίγουν όμω τραπεζικούς λογαριασμούς ή αγοράζουν έγκαιη ιδιοκτησία ή κάνουν οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνουμε ε, μια αρμόδια διοκτική αρχή FIU σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα συντονίσει τη δράση της με τις εθνικές και θέλουμε να ακούσουμε την Επιτροπή για τις ανώνυμες προπληρωμένες πιστοτικές κάρτες ε, γιατί πρέπει να μας πει τι θα κάνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την καταπολέμηση της Θα κάνουμε και τροπολογίες για τις ε, ευθύνες ε, των αυτορυθμιστικών ε, αυτοδιαχειριζόμενων επαγγελμάτων, νομικών επαγγελμάτων και άλλων. Ευχαριστούμε, Μπέρντ. Λούκε. Από το ECR. Δεν έχουμε χρόνο. Ε, συγγνώμη, Πρόεδρε, υπάρχουν κάποιοι που δεν υπερβαίνουν το χρόνο τους και θα πρέπει να το λαμβάνετε υπόψη γιατί οι υπόλοιποι σκιώδεις δεν έχουν χρόνο στη διάθεση. Για να δούμε τι θα κάνετε. Καλά, θα μιλήσω γερμανικά. Ε, ουσιαστικά είμαι υπέρ των προσπαθειών που κάνουν οι συγητές εδώ. Ο στόχος είναι καταπολέμηση του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, να κλείσουν τα παραθυράκια. Έχει γίνει καλή δουλειά, όμως ε, πρέπει να συζητήσουμε και το, η έκθεση επιδέχεται βελτιώσεις. Ε, κυρίως για το μητρό των ε, beneficial ownerships, ε, δηλαδή των οικονομικών φορέων δικαιούχων που θέλουμε να είναι προσβάσιμες στις διοκτικές αρχές αυτά τα μητρώα, αλλά αυτή η διατύπωση που λέει πρέπει να υπάρχει θεμητό συμφέρον. Δεν έχει οριστεί η έννοια όμως, οπότε θα είναι εύκολο να παρακαμφθεί. Και δεν υπάρχει και καμία εγγύηση σε σχέση με τον τρόπο υπεύθυνου ε, χειρισμού των πληροφοριών, των δεδομένων. Ε, τα παραθυράκια που πρέπει να κλείσουμε, ε, ποια είναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει για τα ιδρύματα να καταχωρίζονται εκεί όπου είναι ο τόπος διοίκησής τους, η έδρα διοίκησής τους. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά ιδρύματα και οντότητες που ε, σε εξωχώρια εδάφη έχουν την έδρα τους, ε, τη διοικητική τους έδρα, στην Καραϊβική συγκεκριμένα. Ε, και οπότε για να κλείσουμε αυτά τα παραθυράκια, πιστεύω ότι δεν βελτιώνει την κατάσταση η πρόταση του εισηγητή, διότι λέει η διατύπωση εκεί που είναι η διοικητική έδρα εκεί που ε, ε, προκύπτει η προσθέμενη αξία, εκεί που αναπτύσσεται ε, η εμπορική δραστηριότητα. Θα εξακολουθήσει να υπάρχει το παραθυράκι όμως με αυτή τη διατύπωση. Θα πρέπει να πούμε ότι θα, πρέπει να υπάρχει επίσημη καταχώρηση σε ένα κράτος μέλος αυτού του Ιδρύματος. Το σημαντικό είναι να είναι στα Μητρώα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε μιλάμε για ίδρυμα είτε για τράστε. Δηλαδή εκεί που δραστηριοποιούνται οικονομικά. Επίσης, εξαιρέσεις για όσους δέχονται εκβιασμούς, ε, εκφοβισμό, ε, δωροδοκία ε, ε, ε, ξέρετε ότι για πάρα πολύ πλούσιους ανθρώπους είναι σύνηθες αυτό και είναι τεράστια η τρύπα που αφήνουμε στο νομοθέτημα και θα πρέπει να αποκαλύπτεται η ταυτότητα των beneficiaries, των δικαιούχων για τους ανήλικους ή για τα αμαία άτομα με ειδικές ανάγκες κατά τη γνώμη μου, πρέπει να απαιτούμε τουλάχιστον οι νόμιμοι κυδεμόνες τους ε, να είναι γνωστοί, να είναι γνωστή η ταυτότητά τους, γιατί αλλιώς θα ανοίξουμε ένα παραθυράκι, γιατί αυτά, αυτοί οι ανήλικοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους, οι δικαιούχοι δεν ε, είναι άγνωστοι, δεν γνωρίζουμε την ταυτότητά τους. Ε, σε σχέση με τα ευρωπαϊκά μητρώα υπάρχει και το θέμα της γλώσσας. Είναι η τελευταία παρατηρήση, Πρόεδρε. Ναι, υπερβαίνετε κι εσείς το χρόνο σας, αλλά δεν πειράζει, συνεχίστε. Ε, λοιπόν, ε, ε, σε 24 γλώσσε πρέπει να είναι διαθέσιμε οι πληροφορίε. Και πώ θα υποχρεώσουμε την οντότητα ε, σε ένα άλλο κράτο μέλο ε, να κάνει όλη αυτή την έρευνα σε ξένε γλώσσε, και χρειαζόμαστε μια τυποποίηση ούτω ώστε ακόμη και να είναι σε κάποια άλλη γλώσσα διαθέσιμη πληροφορία να μπορεί τάχιστα να είναι διαθέσιμη. Α, δεν το βρήκατε ούτε σε εύκολο να είστε σύντομο. Ο κύριο Τζάζεκ, πάντοτε σύντομο σωστά. Εσείς δεν έχετε πρόβλημα. Νομίζω πως η πρόταση της Κομισιόν είναι ήδη θετική και το σχέδιο του το δικό μας το ενισχύει. Φυσικά και θέλω να υιοθετηθεί μια φιλόδοξη ε, προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε τις τα εναπομείνοντα παραθυράκια μετά από την υπόθεση Panama Papers, ώστε να καταστεί ακόμα πιο σαφές ότι είναι το σωστό εργαλείο αυτό για να προχωρήσουμε. Τώρα για τις τροπολογίες, το σχέδιο έκθεσης για τον εντοπισμό των, ε, της ιδιοκτησίας δεν νομίζω πως θα πρέπει να αφήσουμε χώρο ώστε να μπορούν να παρακάμψουν αυτή την υποχρέωση οι δικαιούχοι αυτοί και όταν θα υπάρχει μια αφιβολία θα πρέπει να τονίζεται και στην έκθεση και θα μπορούσαμε αυτό να τον ισχύσουμε ακόμη περισσότερο ε, ασκώντας πίεση στην εταιρεία ή στον όμιλο ώστε να κάνει αυτή την καταγραφή απαιτώντα οποιαδήποτε ε, μονάδα να, να έχει μια, να δώσει μια απόδειξη της καταγραφής, της εγγραφής στο Μητρό από τη στιγμή για να μπορεί να ξεκινήσει τις, τις δραστηριότητε της. Επίσης θα πρέπει να είναι δημόσιο αυτό το Μητρό και στηρίζω τις τροπολογίες που περιορίζουν ή πλαισιώνουν τις εξαιρέσεις που μπορεί να κάνουν τα κρατη οι εξαιρέσει θα πρέπει να παραμένουν εξαιρέσει και είμαι ευτυχή που η έκθεση ενισχύει τι διατάξει για τη συνεργασία ανάμεσα στι NFIU και τι αρμόδιε αρχέ και να εστιάσουμε σε αυτή τη συνεργασία και με τρίτε χώρε. Θα ήθελα επίσης να διερευνηθεί δυνατότητα ενός ευρωπαϊκού FIU που θα στήριζε τα εθνικά. Υπό το φως των τελευταίων χωρών ψηλού κινδύνου που προτείνει η Κομισιόν, που είναι πολύ μικρός ο κατάλογος, θα πρέπει να ενισχύσουμε τον κατάλογο των κριτηρίων που χρησιμοποιεί η Κομισιόν για να εντοπίσουμε αυτές τις χώρες. Ο εισηγητής επίσης ε, ήδη προσθέτει ένα παραπάνω κριτήριο και θα πρέπει να διερευνήσουμε αν πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ και επόμενο σκιώδης της ΕΚΟΝ είναι ο Μάρκο Βάλι, FDT. Ναι, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσον αφορά την ομάδα μου, η πρόταση της Κομισιόν για αναθεώρηση της οδηγίας κατά της ανακύκλωσης και η εργασία των συνεισηγητών ακολουθεί την σωστή κατεύθυνση. Στηρίζουμε την εισαγωγή της πρότασης της Κομισιόν ε, ενός δημόσιου μητρώου για τους πραγματικούς δικαιούχους των ομίλων και των εταιριών. Αν και υπάρχει χώρος για βελτίωση θα πρέπει να υποβάλουμε τροπολογίες και εκτιμούμε την προσπάθεια των συνεισηγητών για βελτίωση αυτού του κειμένου ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα ιδιαίτερα μετά από ένα σωρό σκάνδαλα τα οποία αντιμετωπίσαμε και στις αρμόδιες επιτροπές. Θεωρούμε πως είναι απαραίτητο να μειωθεί το κατόφλι ε, το, της μετοχικής συμμετοχής για να μπορούμε να εντοπίσουμε τους πραγματικούς ιδιοκτήτες. Με το κατόφλι που προτείνεται αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα των κινέζικων κουτιών ούτε και το πρόβλημα της ανακύκλωσης και των παράνομων δραστηριοτήτων όπως το γνωρίζουμε. Το κατόφλι θα έπρεπε να είναι πολύ χαμηλότερο, τουλάχιστον το 10%. Θα θέλαμε πολύ δηλαδή να μειωθεί αυτό το κατόφλι και τα όσα προβλέπονται από την πρόταση για τις παθητικές όπως λέγεται μη χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες. Το κατόφλι του 25% είναι δεκτό. Μετά έπειτα όλοι οι όμιλοι θα πρέπει να υποχρεούνται να δώσουν στοιχεία στο να δημοσιεύσουν στοιχεία για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες ε, χωρίς διακρίσεις. Η πρόταση της Κομισιόν ανάμεσα σε εμπορικούς ομίλους και μη και εμπορικούς ε, ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα ως παραθυράκι και μπορεί να υπάρξει εδώ κατάχρηση. Έπειτα, η, το μητρό των πραγματικών ιδιοκτητών, των εταιριών και των ομίλων θα πρέπει να είναι μια βάση δεδομένων δημόσια και διαθέσιμη σε όλους. Θα έπρεπε να απαγορεύεται λοιπόν καταγεγραμμένους να εφαρμόζουν ε, τη μέση αμοιβέ. Θα πρέπει να είναι απόλυτα δημόσια και προσβάσιμη αυτή η βάση. Αυτέ είναι οι τροπολογίε που στηρίζουμε από πλευρά των συνεισηγητών. Δεν χρειάζεται τώρα να σα τι απαριθμίσω. Θα σταματήσω σε αυτά και ελπίζω όντω ότι θα συνεχιστεί αυτή η σπουδαία συνεργασία μεταξύ όλων γιατί υπάρχει καλή βούληση για συνεργασία και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, όπως βλέπετε, αρκετοί από τους κοιόδης δεν είναι εδώ. Και γι' αυτό θα έχουμε χρόνο να δώσουμε ε, το, λόγο και σε άλλους ομιλητές, όπως η κυρία Χολμάγερ. Να, Μπερές. Συγγνώμη, το όνομά σας δεν θυμάμαι. Εντάξει, θα μου πει η γραμματεία. Δύο από την ΕΚΟΝ και δύο από την ΛΥΠΗ. Τι στις Δης. Α, με συγχωρείτε. Δεν σας έχω γνωρίσει. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, δεν σας γνωρίζω. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ τους εισηγητές για την προσπάθεια που έκαναν Ε, προσπάθησαν να έχουν μια συνεκτική ισχυρή θέση. Θέλω να πω κάποια πράγματα για τα καταπιστεύματα και το ποσοστό 25% είναι υπερβολικά υψηλό. Και παρότι για τις παθητικές ε, μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες προτείνει μείωση του ποσοστού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλουμε να μειώσουμε το όριο στο 5% για όλες τις εταιρείες, όπως σε κάποια κράτη-μέλη για το παραθυράκι σε σχέση με τον το διευθυντή. Συμφωνούμε, αλλά θέλουμε να κάνουμε άλλο ένα βήμα, δηλαδή η οντότητα θα πρέπει να πάυσει ε, την οικονομική συναλλαγή εάν δεν υπάρχει, ε, είναι γνωστή η ταυτότητα του δικαιούχου, δεν υπάρχει beneficial ownership. Αν δεν θέλει να κοινοποιήσει τα στοιχεία, δηλαδή. Για το Μητρό πλήρη πρόσβαση ζητάμε, χωρίς ε, καμία δυνατότητα εξαίρεσης. Για την πράξη εξουσιοδότηση η Τζούντιθ το είπε. Ελπίζω ε, να βρούμε υποστήριξη από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες και να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν αρκεί αυτό, χρειαζόμαστε πλήρη κατάλογο. Ευχαριστούμε. Ο Ντένις Τεγιόγκ έχει γραφτεί ως Α, είχαμε τον Ντένις Τεγιόγκ αντί για σας, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Η ε, κυρία Χολμάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπροσωπώ τον Σκιώδη ε, εισηγητή ε, και δεν ε, υπήρχε μετάφραση, διερμηνία γι' αυτόν και είναι ατυχές. Μιλάει η συγγήτρια γερμανικά και αγγλικά, αλλά μιλάει τεχνική ορολογία και... Και δεν είναι φυσιολογικό να μην έχει διερμηνία η σκιώδη συζητήτρια, γιατί... Ή... Σκιώδη γιατί αλλιώς ε, δεν μπορεί να εκφράσει τεχνικές απόψεις. Λοιπόν, ε, τα εικονικά νομίσματα, bitcoins, ε, Ε, ε, είναι το ε, σημαντικότερο σημείο μέσα στα, στην οδηγία και θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί γιατί στο σκοτεινό δίκτυο, το dark web, είναι από τα πιο συχνά φαινόμενα για την τρομοκρατία και τις διοκτικές αρχές ε, υπηρεσία πληροφοριών, αστυνομία, ε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επαλήθευσης ελέγχου ε, για να υπάρχουν εντατικοποιημένοι ελέγχοι και δυνατότητα συλλογής και συγκέντρωσης των απαραίτητων πληροφοριών. Να προσθέσω και εγώ κάτι που θεωρώ σημαντικό. Due diligence, θέως επιμελητία. Ε, ε, συγγνώμη, επιμέλεια. Ε, μην ξεχνάμε ότι δεν πρόκειται για μεγάλες ε, συναλλαγές, ε, για το πετρέλαιο, για τα διαμάδια, για το χρυσό, για τα χρηματιστήρια αγαθών. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται φυσιολογικοί διαβλοί και οι πολιτές δεν χρειάζεται να κοινοποιήσουν την ταυτότητά τους. Είναι ιδιαίτερα προβληματικό και Χαίρομαι πάρα πολύ ε, που μου δώσατε το λόγο και ο κύριος Δράντεφ ε, στέλνει και πολλούς χαιρετισμού και ελπίζει να είναι εδώ την επόμενη φορά. Ε, ε, ναι, πολύ, πολύ λογικό αυτό που είπατε και έγινε δεκτό. Το σημειώσαμε τα, αυτό που είπατε περί διερμηνία. Ήταν που οργανώθηκε τελευταία στιγμή η συνεδρίαση. Ρομπέρτα, σε πειράζει να πάρουμε κάποιον από την ΕΚΟΝ και μετά. Mm. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους εισηγητές για την πάρα πολύ καλή βάση εργασίας που μας ε, προτείνουν. Θα ήθελα λίγο να επιμείνω ε, στα δύο άκρα αυτής της αλυσίδας. Συμφωνώ σε πολλά σημεία με την κυρία Χολμάιερ για τα εικονικά νομίσματα και τα bitcoin και τον τρόπο με τον οποίο η Κεντρική Τράπεζα μας προειδοποιεί για όλο αυτό το διακύβευμα των εικονικών νομισμάτων. Στην ΕΚΟΝ ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Τρέχει μια έκθεση τώρα για το FinTech, αλλά δεν μπορούμε να ε, παραβλέψουμε και από αυτή τη σκοπιά τα εικονικά νομίσματα. Εξού και ξανανοίγει αυτή η οδηγία η MLD για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτό το θέμα μας έχει απασχολήσει από την αρχή και μπορεί να μας ενδιαφέρει και στη συνέχεια. Τώρα στο άλλο άκρο της αλυσίδας είναι το θέμα του κατοφλίου για τις προπληρωμένες κάρτες. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Ευχαριστώ τον εισηγητή που ε, η υποτριπλασίασε το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, αλλά θα πρέπει εμείς να πάμε ακόμα παραπέρα. Ακούμε συχνά ένα επιχείρημα που λέει, μα οι προπληρωμένες κάρτες, εάν τις ανοιχνεύουμε, αυτό είναι εις βάρος εκείνων που είναι εκτός του τραπεζικού ή του νομισματικού κυκλώματος. Δεν ευσταθεί αυτό το επιχείρημα, γιατί η προπληρωμένη κάρτα είναι πληρωμένη. Δεν τίθεται θέμα ε, αν έχεις πρόσβαση στα χρήματα στις πιστώσεις. Δεν σε ρωτάει κανείς πόθεν έσχες, πού τα βρήκες και πλήρωσες αυτή την κάρτα και την αγόρασες. Αν θέλουμε όμως να τις ανοιχνεύουμε με τρόπο σοβαρό στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δεν υπάρχει λόγος να φτάσουμε στο μηδέν. Καμία σχέση δεν έχει αν έχει λογαριασμό σε τράπεζα ή όχι. Και ένα τελευταίο θέμα είναι ε, το θέμα αυτό των trusts. Ε, είναι κάτι που επανέρχεται συνέχεια και νομίζω ότι υπάρχει χώρος για πρόοδο. Και μέσω των τροπολογιών ελπίζω να βελτιώσουμε την περαιτέρω την πρόταση. Ευχαριστώ, Περβάνς. Η κυρία Μέτσολα, τελευταία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να κάνω μια γενική παρατήρηση επί της αρχής. Το σκάνδαλο των Χαρτιών του Παναμά έχει εκθέσει τη διεφθαρμένη ε, διαδραστηριότητα ξεπλήματος μαύρου χρήματο σε σχεδόν βιομηχανικό ε, επίπεδο και έχει δείξει ε, τη συνεργασία των κρατών μελών για αυτά τα πράγματα και την ανικανότητά τους να κάνουν οτιδήποτε. Όταν πρόκειται για ξέπλυμα χρήματο, θα πρέπει να προσέχουμε να μην βιαστούμε για να μην κάνουμε λάθος. Κατά τη γνώμη μου, εγώ θα πρόσεχα πολύ θα έπρεπε να προσέξουμε πολύ μην κάνουμε δυσανάλογη νομική, μάλλον νομοθετική απάντηση που μπορεί να ε, παρέμβει στην κυριαρχία των κρατών σε θέματα φορολογία υπό την, το πρόσχημα της, ε, του, κυνη, του κυνηγιού του ξεπλήματο ε, ε, μαύρου χρήματο. Για τη Μάλτα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτέ οι νομοθεσίε δεν θα επιβαρύνουν οικονομίε όπω η δική μα υπερβολικά. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε εδώ είναι η καταχρηστική παράνομη δραστηριότητα δηλαδή το ξέπλυμα χρήματο και όχι η φορολογική ανταγωνιστικότητα του κράτους. Ευχαριστώ κυρία Μετσόλα και τώρα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές και τους κοιόδες για την συμβολή τους και για την εργασία τους αλλά και για την συνεργασία ανάμεσα στις επιτροπές που είναι εξαιρετική. Θα ζητήσω τώρα από τον συνεισηγητή μου συμπρόεδρο μάλλον εννοεί ο πρόεδρος, ε, να μας πει ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Την Κομισιόν να ακούσουμε. Όχι. Την Κομισιόν δεν θέλει, δεν θέλει. Καλά, δεν πειράζει. Κυρία Σαρτζεντίνη, έχετε κάτι διαδικαστικό. Ναι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θα κάνουμε με τις κατεξουσιοδότηση πράξη. Γιατί νομίζω πως έμεινε ναι, αλλά δεν άκουσα όλε τι, όλες τις ομάδες. Α, άλλαξε την γνώμη της τώρα η Κομισιόν. Ναι, παρακαλώ, ναι, πείτε μας, αλλά σύντομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Δεν ήθελα να πάρω το λόγο γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ε, είναι πολύ καλή η συζήτηση σήμερα. Είναι ένα, ένα σημείο κίνησης ε, η πρότασή μας. Θα βρούμε τρόπους για να βελτιώσουμε το κείμενο. Να κάνω μια παρατήρηση ίσως ε, στη συνέχεια για, για τον κατάλογο των τρίτων χωρών, αλλά πρώτα να, να σας ακούσω ή τώρα. Α, τώρα. Λοιπόν, για να μην δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση ότι κάνουμε copy-paste ε, για τους καταλόγους της ΦΑΤΦΑ, η οδηγία για την νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων μας επιτρέπει να έχουμε μια αυτόνομη διαδικασία και προσδιορισμό κριτηρίων για να αποτιμήσουμε τις, ε, την επικινδυνότητα των τρίτων χωρών. Φυσικά κοιτάζουμε τι κάνουν οι διεθνείς οργανισμοί για την αξιολόγηση και αυτά που κάνει η ΦΑΤΦΑ ε, μας ενδιαφέρουν ε, και ε, τα εξετάζουμε, αλλά δεν είναι μοναδική πηγή που χρησιμοποιούμε. Δούμε Υπάρχουν ε, πάντως ε, ε, ελλείψεις και σταδιακού χαρακτήρα και έχουν ληφθεί μέτρα για για τα χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις. Γιατί Ε, ε, ήδη εγγύσει την εξέταση και θα συνεχίσουμε για τις υπόλοιπες τρίτες χώρες. Ευχαριστούμε. Ο θα μας μιλήσει για το χρονοδιάγραμμα, πώς θα συνεχίσουμε. Δεν βλέπω να υπάρχουν μεγαλύτερες ε, φιλοδοξίες, ε, ξέρετε. Όλοι συζητάνε για τον Παναμά, εκτός από εσά ε, για απευθύνομαι στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα δούμε πώς θα αντιδράσουν και οι άλλοι. Οι συντονιστές ε, ίσως εκπονήσουν σχέδιο ψηφίσματος για το εργοποιημένο πράγμα κατα, εξουσιοδότηση. Σήμερα στις 12 είναι η προθεσμία και συνεχίζεται η γραπτή διαδικασία διαβούλευσης. Ένας μήνας είναι η κανονική περίοδος εξέτασης και θα στείλουμε επιστολή για παράταση κατά ένα μήνα. Μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2017 θα τρέξει η προθεσμία και τι σημαίνει αυτό ότι το σχέδιο ψηφίσματος πρέπει να πάει στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο 2017 και η Μεκτή Επιτροπή πρέπει να το Δεκέμβρη να ε, ψηφίσει για το σχέδιο, Σε 8 μάλλον θα συνεδριάσουμε. Το σχέδιο μπορεί να κυκλοφορήσει και αύριο, μόνο στα αγγλικά. Ε, βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών για την εξέταση της ΕΚΟΝ, ο εισηγητής ε, για την αρχική πράξη θα είναι ο συντονιστής, ε, ε, η σκιώδης, ε, μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 11 η ώρα θα μπορέσουμε να καταθέσουμε ε, τροπολογίες για το σχέδιο αυτό, αλλά πάλι μόνο στα αγγλικά. Αυτά! Και σας ευχαριστώ που ήρθατε όλοι τόσο νωρίς. Να έχετε μια ε, καλή και ευχάριστη μέρα εργασίας.